Allora abbiamo proceduto alla eh, Ψηφίσαμε ο υποψήφιος για το ηλεκτρικό συνέδριο από την Αυστρία, ο κύριος Φόγκεμπάουερ, πήρε 13 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά, 6 αποχές. Με πλειοψηφία λοιπόν ε, ψήφος θετική. Και ερχόμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα του προπλησμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη-μέλη. Ψηφοφορία. Ο συνάδελφος Μαρινέσκο θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Το νόημα αυτής της έκθεσης κατά τη γνώμη μου είναι να ζητήσουμε από την Επίτροπη ε, και από το ελεγκτικό συνέδριο, διότι ετοιμάζουν νέες αξιολογήσεις αυτού του προγράμματος, να τους ζητή, ε, θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις και να έχουμε τις απαντήσεις στο μέλλον, για, στη μελλοντική έκθεση αυτή η εισήγηση δεν προτίθεται να διακόψει ή να παρατείνει τη χρηματοδότηση, αλλά προτίθεται να βρει απαντήσεις για να δει αν χρειάζονται ακόμα κονδύλια ε, για το πρόγραμμα αυτό ή όχι και πώς ε, θα ε, ξοδευτούν τα χρήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Έναρξη ψηφοφορίας. La votazione è Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Έναρξη. 6. Απορρίπτεται. 12. Έναρξη. Πέρασε. Μετά θα το κάνουμε όχι με τις κάρτες, αλλά με τα διενάτες χειρός. Αν συμφωνείτε. Η 12 εγκρίθηκε ή όχι. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία της τροπολογίας 12, έναρξη. Ποιος είναι υπέρ με τα χέρια. Κατά. Συγγνώμη, καλύτερα ηλεκτρονικά. Γιατί αν μετράμε τα χέρια, όχι. Μην με μπερδεύετε με τις κάρτες. 12 ψηφίζουμε με τις κάρτες, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 έναρξη και λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 έναρξη και λήξη. Απορρίπτεται. Εκεί τρία Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεκαεννέα, Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 21 έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 22 έναρξη αποσύρεται 23 έναρξη λήξη εγκρίνεται 24 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παραθμόν 4. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 28. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται 31 έναρξη λήξη εγκρίνεται 32 έναρξη λήξη εγκρίνεται 34 έναρξη λήξη εγκρίνεται 35. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 36. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 37. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 38. Έναρξη. λήξη απορρίπτεται 39 έναρξη λήξη εγκρίνεται 40 έναρξη λήξη απορρίπτεται 41 έναρξη λήξη εγκρίνεται 42 έναρξη λήξη απορρίπτεται 43 έναρξη λήξη απορρίπτεται 44 και 45 έναρξη Λήξη. Απορρίπτεται. 46. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 47. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 48. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 49. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμόν 6. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 52. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 53. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 54. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 56. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπεραθμόν 7. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 63 έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 64 έναρξη λήξη εγκρίνεται 65 έναρξη λήξη εγκρίνεται 66 έναρξη λήξη εγκρίνεται 67 έναρξη λήξη εγκρίνεται 68 έναρξη λήξη εγκρίνεται 69 έναρξη λήξη εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 1 έναρξη λήξη εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 2 έναρξη λήξη Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογία της Ήτρα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της ήθρα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 Ήτρε δεύτερο τμήμα έναρξη λήξη εγκρίνεται Τροπολογία 8 έναρξη λήξη εγκρίνεται Τροπολογία 9 έναρξη λήξη απορρίπτεται Αιτιολογική σκέψη Γ, τη Ήτρε. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο, ε, το, το ψήφισμα με τις αλλαγές. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται με 22 ψήφους κατά, κανένας, καμία ψήφο κατά και μία αποχή. 23 ψήφους, 22 ψήφους υπέρ. Συγχαίρουμε τον εισηγητή και προχωρούμε. Με το σημείο 6 το μέλλον της δημοσιονομικής στήριξης της Ένωσης της αναπτυσσόμενες χώρες, εισηγητής του συνάδελφου ΣΤΑΣ στον οποίο και δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ένα έγγραφο στα χέρια σας, ε, το υπαριθμό 6 που είναι το σχέδιο γνωμοδότησης μου προς την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πέρα από αυτό έχω διανύμει και ένα άλλο έγγραφο που είναι πιο διευρυμένο με τις τροπολογίες του εισηγητού. Στα αγγλικά το λέει αυτό. Γιατί το έκανα αυτό. Μια τέτοια γνωμοδότηση είναι πάντα πολύ περιορισμένη. Είχα ε, 2.000 χαρακτήρες για να πω στην πρώτη πρότασή μου τι θέλω να κάνω για την υποστήριξη του προπολογισμού και για την πράσινη βίβλο και δεν έφταναν καθόλου, όπως καταλαβαίνετε, οι 2.000 χαρακτηρίες για να κάνω εκτενή γνωμοδότηση. Οπότε σε πρώτη φάση έχω γράψει 7 συστάσεις και θα ήθελα να τις συμπληρώσω με τις προτάσεις ε, στο έγγραφο που σας μοίρασα και που είναι με τους ε, έντονους χαρακτήρες. Θα έρθω και σε επαφή με τους συντάκτες του τροπολογιού, αν θέλουν να τις υποβάλουμε από κοινού. Η δημοσιονομική στήριξη στον κόσμο της αναπτυξιακής βοήθειας τι σημαίνει. Αν ακούσετε τους ενδιαφερομένους και εκείνους που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, όλο και περισσότερο είναι ένα μέσο αυτό που χρησιμοποιείται και γενικότερα ο κλάδος το αξιολογεί αρκετά θετικά. Στην πρώτη μου λοιπόν σύσταση λέω αναγνωρίζει ότι είναι καλό μέσο ανάπτυξης και αποτελεσματικό, δεδομένου ότι σέβεται απόλυτα κάποιες ε, ουσιαστικές αναπτυξιαρχές αρχές, δηλαδή το να έχει κάνει ο δικαιούχος κτήμα του αυτή την υπόθεση, το ownership που ε, είναι της μόδας όρος και ε, η τεχνική αυτή ε, συνδέεται και με χαμηλότερα ή χαμηλά ε, κόστη ε, συναλλαγών. Δεν είναι όμως η μόνη λύση ούτε πανάκια για την επίλυση όλων των προβλημάτων παγκοσμίως. Επόμενη σύσταση ή παράγραφος. Δεύτερη. θα πρέπει να διασφαλίζεται ε, ο στόχος της συμπληρωματικότητας με τα εθνικά προγράμματα. Μια ανεπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να είναι ξεκάρφωτη από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Και επίση η δημοσιονομική ενίσχυση θα πρέπει να ε, συσχετίζεται κάπως και να συντονίζεται και να συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες. Και πάντα ε, σε αρμονία ή σε συνοχή με άλλη υποστήριξη που δίνουν άλλοι δωρητές δεν είναι κάτι το αποσπασματικό, το ξεκομμένο, ένα νησί ας πούμε στο πουθενά. Επιπλέον θα πρέπει η βοήθεια στον προπολογισμό να είναι ε, προσθετική. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι Βέλγος και έχουμε ισχυρή σχέση με την πρώην επικία, απικία μας στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και αν δει κανεί πώς λειτουργεί εκεί το καθεστώς και αρκετά περιορισμένο ε, προεπολογισμό. κάθε ας πούμε ο πρόεδρος Καμπίλα και λέει αφού θα πάρω αναπτυξιακή βοήθεια για τη δημόσια υγεία, ε, δεν θα γράψω κονδύλι στον προπολογισμό μου. Αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να είναι ε, η δημοσιονομική ενίσχυση ε, επιπλέον των όσων προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση της χώρας σε ένα κλάδο. Όχι να το υποκαθιστά, αλλά να το συμπληρώνει με τον κατάλληλο τρόπο. Κάτι άλλο που δεν λέει η πρότασή μου και θα το κάνω ως τροπολογία και θα το βρείτε στο καινούργιο έγγραφο με τους έντονους χαρακτήρες το 2α δηλαδή. Ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ευθυγραμμίσει τον προγραμματισμό της και το σχεδιασμό με τις προετοιμασίες και την τεκμηρίωση Δηλαδή να γίνει με έναν τρόπο συντονισμένο, αυτό το λένε streamline στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επαρκές προσωπικό εκπαιδευμένο που να γνωρίζει τα θέματα αυτή της δημοσιονομικής διαχείρισης και μεταξύ άλλων ιδιωτήτων και ικανοτήτων και προσόντων που θα πρέπει να έχει το προσωπικό αυτό θα πρέπει να ξέρει ότι είναι διαφορετική τεχνική. Ε, χρειάζεται πιο ε, αναλυτικές ε, ικανότητες ή περισσότερες αναλυτικές ικανότητες, σε πάση περιπτώσει, από άλλα projects ή άλλα έργα που χρηματοδοτούμε. Είναι κάτι το διαφορετικό. η τρίτη παράγραφος, στο μεταξύ τέταρτη, γιατί έχουμε βάλει και το 2α, θα πρέπει οι στόχοι να είναι διατυπωμένοι με τέτοιο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή τη μέτρηση, λέω, της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και να λαμβάνει δεδόντως υπόψη τις ανάγκες προτεραιότητας της δικαιούχου χώρας. Τέταρτη σύσταση. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην αξιολόγηση των ελέγχων Μάλλον να το πω αλλιώς. διορθώνει ο μιλητής γιατί λάθος το διατύπωσε. Θα πρέπει να να εξελιχθούμε, να ξεφύγουμε από τον έλεγχο των εισρώων, αλλά ε, να πάμε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων με δείκτες, να μετράμε ε, την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης ε, για να δούμε αν τρέχουν σωστά τα προγράμματα. Πέμπτον, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στους κινδύνους διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, γιατί πολύ συχνά δεν είναι πολύ ισχυρή η διοίκηση της χώρας από πλευράς του δημοσίου κάθε φορά στις χώρες που επεμβαίνουμε και θα πρέπει να έχουμε συστήματα διαχείρισης του κινδύνου αποτελεσματικά. 5α ε, τώρα νέο, τροπολογία στο νέο κείμενο, εκφράζω κάποια ανησυχία. Το ε, ελεγκτικό συνέδριο σε πολλές ειδικέ του εκθέσεις απεφάθηκε για τη δημοσιονομική ενίσχυση και έχει κάνει και μια σύντομη έρευνα. Και από όλη αυτή τη μελέτη και την έρευνα δείχνει ότι όλο και περισσότερο έχουμε σφάλματα μη μετρήσιμα που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στη δημοσιονομική στήριξη, στη μακροοικονομική βοήθεια και στη παράγραφο 5β τροπολογία ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυάται ότι οι αντιπροσωπείες ε, που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα στις δικαιούχες χώρες συστηματικά να κάνουν εκθέσεις διαρθρωτικές και τυποποιημένες για την πρόοδο που επιτελείται και που έχει σημειωθεί. Με βάση κριτήρια τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Ανησυχώ εγώ, όταν δίνει ενίσχυση στον προπολογισμό σε κάποια χώρα πρέπει να έχει κάποια κριτήρια, κάποια συμφωνία για να μπορεί να τα μετρά όλα αυτά και να τα αξιολογήσει εκ των υστέρων. Η αρχική μου παράγραφος 6 καλεί και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στις δικαιούχες χώρες. Πώς καταπολεμάται η διαφθορά, τι χρειάζεται εκεί. Καλό διάλογο και ισχυρό διάλογο με τις κρατικές αρχές να υπάρχει δυνατότητα οικοδόμησης ε, των θεσμών, των δυνατοτήτων και να φροντίζουμε για μηχανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς και υπευθυνότητας. Η παράγραφος 7 ε, του αρχικού μου κειμένου ε, ζητάει από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από την Κοινωνία των Πολιτών και τις τοπικές αρχές των εταίρων χωρών να συμμετέχουν. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι τον αφορούν αυτά τα θέματα, είπαμε να τα αισθενιστεί, να τα κάνει κτήμα του και να τα υλοποιεί. Και ένα τελευταίο, τελευταία παράγραφος, 7α στο νέο κείμενο, πάλι με έντονους χαρακτήρες, εκεί λέγω, κοιτάξτε, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, στον αντίστοιχο κανονισμό, που διέπει αυτή τη ε, δημοσιονομική βοήθεια και την περιγράφει, έχουμε το άρθρο 25β, το οποίο ορίζει, και θα το διαβάσω στα αγγλικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει συστηματικά να χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που να βασίζεται σε δείκτες αποτελεσμάτων και επιδόσεων και να ορίσει σαφώς όσο και να ελέγχει ε, την ε, και να υποστηρίζει τις προσπάθειες των εταίρων χωρών για να αναπτύξουν κοινοβουλευτικό έλεγχο και ικανότητες λογιστικού ελέγχου και να αυξήσουν τη διαφάνεια και την πρόσβαση του κοινού στην ενημέρωση. Αυτό ισχύει για την επίσημη ε, αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μεταφερθεί ως κατευθυντήρια γραμμή, ως ε, Ηρμός και στην υποστήριξη τη δημοσιονομική. Το λέω και στην τροπολογία μου. Ε, μόνο τα τεχνικά κριτήρια του άρθρου 61 εδάφιο 2 της Συμφωνίας Κοτονού δεν αρκούν ε, ε, αυτές οι τεχνικές ρυθμίσεις και μόνο. Χρειάζεται να μεταφέρουμε και αυτή την παράγραφο να ισχύει και για τη δημοσιονομική βοήθεια πέρα από την εκεί. Αυτά, αν συμφωνείτε, θα τα υποβάλω ως τροπολογίες του εισηγητού και με τις άλλες τροπολογίες των διαφόρων πολιτικών ομάδων για να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας. Είναι ευρύτερο από αυτό που είχα γράψει αρχικά λόγω του περιορισμού 2.000 χαρακτήρες, κορσές και καλό θα είναι να επιταχύνουμε γιατί στις 28 Μαρτίου πρέπει να ψηφίσουμε γιατί τόσο νωρίς η ε, Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας Στι 11 Απριλίου ψηφίζεται η δική της έκθεση και ήταν ο μόνος τρόπος να επηρεάσουμε και εμεί και να δώσουμε τη δική μας γνώμη στην Επιτροπή αυτή με σωστό τρόπο. Για να ληφθούν και αυτά που θα πούμε υπόψη. Και νομίζω τον Ιούνιο θα πάει αυτό στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια. Ακούω με χαρά όλε σας τι παρατηρήσει τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ το λόγο αν θέλουν στην Κομισιόν και το Ελληνικό Συνέδριο. Αν θέλετε να μιλήσετε. Δεν είμαι το υπεύθυνο μέλος, αλλά θα ήθελα να πω ότι αφού παρακολούθησα τις προτάσεις και τις τροπολογίες. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ καλό να, να βελτιώσουμε την δημοσιονομική ε, στήριξη πάνω σε αυτή τη βάση και να έχουμε συμβάσεις ε, με τις χώρες, τα κράτη, τις κυβερνήσεις, τους συμμετέχοντες, ακολουθώντας τις γραμμές της εισήγησης και των τροπολογιών. Νομίζω ότι τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου θα μπορούν να είναι ικανοποιημένα για αυτήν την περαιτέρω βελτίωση. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Επιτροπή ενθαρρύνεται από αυτές τις προτάσεις που προσδιορίζουν τους τομείς όπου η Επιτροπή πιστεύει ότι παρόλο που έχει δεσμευθεί ε, για το θέμα αυτό μπορεί να βελτιώσει ε, την δραστηριότητα αυτή στο μέλλον. Παραμπτός χάρη στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ε, που είναι αυστηρή αλλά που γίνονται ακόμα τώρα πιο δομημένοι η Επιτροπή άρχισε να αναθεωρεί το πλαίσιο για την αξιολόγηση κινδύνων για να είναι πιο συνεκτικό και να χρησιμοποιείται πιο συστηματικά παντού. Πρόκειται, λοιπόν, ε, ακολουθούμε λοιπόν την ίδια οδό, τον ίδιο προσανατολισμό. Η Επιτροπή πάντοτε ε, έχει δεσμευθεί, ε, ακολουθεί την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Υπάρχουν προκλήσεις για ορισμένες αδυναμίες των δικαιούχων χωρών, γι' αυτό πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα, τα συστήματα αναφοράς και μπορούν πάρα πολλοί πρόοδοι να επιφέρουν περισσότερη αξιοπιστία. Ως τελευταίο σημείο σχετικά με τον ε, συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών πρόκειται και αυτός ένας τομέας πάρα πολύ σημαντικός. Η Κομισιό έχει δεσμευθεί μαζί με τα κράτη-μέλη για μια ε, ε, προσέγγιση συντονισμού μετά την απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης του 2009. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε αυτό το σύστημα και θα σκεφτούμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλει να μιλήσει κανένα συνάδελφο. Κανεί. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 7. Έρχο ε, δημοσίων διαχείριση και Έρχο των οργανισμών. Σάφο Σταυρακάκη, ηγητή, έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις εκθέσεις των διαφόρων οργανισμών και δραστηριοτήτων είναι να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα μαζί ως ε, ένα σημείο. Πρωτού μπούμε στις λεπτομέρειες ε, του θέματος, η απαλλαγή των οργανισμών για το 2009, θα ήθελα να πω ότι είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύει ακράδαντα ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν για προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως η Επιτροπή μας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα ε, χρήματα αυτά ξοδεύονται με τρόπο κανονικό, με τρόπο διαφανή ε, και νόμιμο. Και αν ε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν, δεν ξοδεύονται με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να ζητήσουμε διορθωτικές πράξεις. Έχουμε ε, τις ε, οριζόντιες παρεμβάσεις των οργανισμών και τις ε, κοινέ δραστηριότητες. Νομίζω ότι είναι πλήρης η παρουσίαση όλων των τομέων δραστηριότητας των οργανισμών μεμονωμένα και από κοινού. Το σχέδιο έκθεση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που σχετίζονται με την δημοσιονομική διαχείριση και τις μεταφορές ε, και τις καταργήσεις ορισμένων πιστώσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στον προϋπολογισμό ε, και ακολουθούν την αρχή του ενιαυσίου. Εάν η φύση των προγραμμάτων ε, ε, θέτει ένα αμφιβόλο και αμφισβητεί αυτή η αρχή, θα πρέπει να δούμε πώς πληρέστερα θα εφαρμόσουμε αυτήν την αρχή. Έχουμε τους οργανισμούς οι οποίοι συχνά έχουν ψηλή ταμιακή ε, δυνατότητα. Ε, οι αδυναμίες στην διαδικασία δημοσίων συμβάσεων πρέπει να ενισχύσουν τους ελέγχους του εσωτερικού ούτως ώστε οι συμβάσεις και οι δημόσιοι διαγωνισμοί, οι διαδικασίες τους να εφαρμόζονται αυστηρά ε, και θα πρέπει οι αδυναμίες ως προς τις επιδοτήσεις να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι κοινό σχετίζεται με ορισμένες αδυναμίες σχετικά με ε, τον διορισμό του προσωπικού που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διαφάνεια αυτών των διαδικασιών. Όπως είπα στην αρχή, οι οργανισμοί πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγγυώνται πλήρως την ανεξαρτησία ε, του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων και να, τους ενθυ... και να ενθαρρυνθούν να ενισχύσουν τους ελέγχους για το θέμα αυτό κάλεσα το, το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει μια ενδελεχή ανάλυση ε, της προσέγγισης ε, διαχείρισης των καταστάσεων όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, παράγραφος 15 της έκθεσης. Σχετικά με τα ως συστήματα ελέγχου των οργανισμών είναι σημαντικό οι διευθυντέ ε, κάθε, κάθε οργανισμού να περιλαμβάνουν ε, στις εκθέσεις τους ε, εκθέσεις για την διαχείριση των χρημάτων και συστάσεις και τις δράσεις που λήφθηκαν κατόπιν των συστάσεων. Θα ήθελα να χαιρετήσω από την άποψη αυτή την πρωτοβουλία της Frontex να προωθήσει την εναρμονισμένη δομή ε, για ε, να ζητήσει την ε, απαλλαγή και, να, και το προτείνει αυτό για όλους τους οργανισμούς. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους οργανισμούς να τυποποιήσουν τις δομές τους σύμφωνα με την μορφή, με το σχήμα που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και να περιλάβουν τις δραστηριότητες που θέτουν προκλήσεις, τις, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και τα συμπεράσματα για το οικονομικό έτος. Η τυποποιημένη μορφή μπορεί να δώσει μια σαφή εικόνα σχετικά με την κατάσταση των οργανισμών. Τελευταίο θέμα, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σχετικά με την γενική εισήγηση, θα ήθελα να τονίσω την σημασία των πολιετών προγραμμάτων δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στον οργανισμό να προγραμματίσει καλύτερα τις δραστηριότητες τους και την, να κάνει ανάλυση κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων για κάθε δραστηριότητα και να κάνει διευθετήσεις για την στρατηγική υλοποίηση ούτω ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Σχετικά με τις εκθέσεις των μεμονωμένων δραστηριοτήτων και από κοινού δραστηριοτήτων. Όπως θα δείτε στο φάκελο σας ε, προτείνω απαλλαγή για όλους εκτός από τρεις. Οι δύο οργανισμοί, ε, Ευρωπαϊκή ως Οργανισμός Φαρμάκων, και ε, επίσης την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, την ΣΥΠΟΛ, που έχουν λάβει μια γνωμοδότηση χαρακτηρισμένη από την Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρατόμ σχετικά με αυτές ε, τους τρεις οργανισμούς ε, ζητώ ε, αναβολή της απαλλαγής. Εν συντομία, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, δεν έχω πολλά να προσθέσω για την Ακαδημία, διότι ξέρουμε ότι Έχουμε αφιερώσει σε, προηγούμενες, σε προηγούμενη συνεδρίαση δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως θα δείτε από το σχέδιο έκθεσής μου, υπάρχουν προβλήματα με την διαχείριση των διαδικασιών για δημόσιες συμβάσεις ε, σχετικά με την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την στρατολόγηση του προσωπικού στην παράγραφο 1 και 2 του σχεδίου έκθεσης γενικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι καλά οργανωμένος και λειτουργεί καλά, αλλά ωστόσο για έναν οργανισμό αυτής της σημασίας νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες που εφαρμόζονται. Θα ήθελα να επωφεληθώ της παρουσίας του κύριου Πότ σήμερα και να του ζητήσω να ενημερώσει την Επιτροπή μας για τα μέτρα που ελήφθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, ούτως ώστε να, υπάρχουν, να υπάρχει ανεξαρτησία των εμπειρογνωμών και τα προβλήματα σχετικά με τον διορισμό που προσωπικό, όπως είπα, πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο λόγος του αιτήματό μας, μας να ελέγξουμε με το εσωτερικό έλεγχο και να δώσουμε ε, τα αποτελέσματα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 22. Σχετικά με την Ευρατόμ, εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο οργανισμός υποτίθεται ότι έχει οικονομική αυτονομία, αλλά αυτή δεν είναι η περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που ασχολείται με όλα. Είναι αλήθεια ότι η Ευρατόμ υπάρχει από το 1958 και μόνο το 2008 άλλαξε το καθεστώς του οργανισμού και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Σία, μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι μαζί μας σήμερα να μας ενημερώσει για την κατάσταση σχετικά με την Ευρατόμ ε, και επίσης τον Διευθυντή της Ευρατόμ ε, που είναι παρόν για να μας πει ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να ξεβρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Σχετικά με τις μικτές δραστηριότητες, όσον αφορά τις κοινέ δραστηριότητες, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρίσκονται σε παιδική ηλικία και αντιμετωπίζουν ε, αυτά τα τυποποιημένα προβλήματα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις μας, τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ούτω ώστε να μπορέσουν ε, να προχωρήσουν, ε, να προοδεύσουν από αυτήν την αρχική φάση και να μην παρουσιάζουν προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ο οποίος ασχολήθηκε με τα σημεία 7 ως 34 του, της ημερήσιας διάταξης. Τώρα δίνω τον λόγο στους διάφορους συναδέλφους. Ο κύριος Τζαμπράντη. Κύριε Μπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σταυρακάκη. Εξαιρετική η παρουσίασή του Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλα όσα είπε και θα ήθελα να προσθέσω μερικά και από πλευρά μου. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια γνωρίσαμε εκρηκτική ανάπτυξη ε, στον αριθμό των agencies, των εξωτερικών οργανισμών και αυτό οδηγεί σε προβλήματα, τα είπε και ο εισηγητής. Πόσα απομεινάρια έχουμε και μεταφορές, τα carry-overs τα λεγόμενα, ας πούμε, 80% στον οργανισμό ε, για την αεροπορία το 2009. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα και έχει να κάνει και με τον πολλαπλασιασμό των οργανισμών. Ε, με εκπλήσει βέβαια αυτό, αλλά ε, ακούμε όλο και περισσότερη κριτική προς τους οργανισμούς αυτούς έτσι ώστε με αποτέλεσμα οι καλοί οργανισμοί ας πούμε, του περιβάλλοντος όπως είπε και ο κύριος Σταυρακάκης πληρώνουν τα σπασμένα κάποιων άλλων οργανισμών που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά και αυτό διαδίδεται έτσι και επηρεάζει και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Έχουμε 7 τέτοιους οργανισμούς που έχουν ε, ως αντικείμενο ε, στη συλλογή στοιχείων. Εκεί εργάζονται 530 εργαζόμενοι συνολικά με ένα προπολογισμό 120 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει όλοι αυτοί οι οργανισμοί να είναι ανεξάρτητοι για να μαζεύουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα συνενώσεις, τίποτα συγχωνεύσεις. Και η διοργανική ομάδα καθώς επίσης και μέλη, όπου συμμετέχουν μάλλον μέλη και της δικής μας Επιτροπής, καλό θα είναι να ασχοληθεί πιο εντατικά και να εσκύψει αυτό το θέμα και θα ήθελα περισσότερη ενημέρωση από την ομάδα εργασίας. Καλό είναι να ρίξουμε μια πιο κριτική ματιά και στον αριθμό των οργανισμών αυτών και πραγματικά μας χρειάζονται όλοι αυτοί. Φέτος θα κάνει μια πρόταση, μια έκθεση στο ελεγκτικό συνέδριο, την οποία περιμένω για, με ανυπομονησία και μεγάλη προσμονή για τη ΣΕΠΟΛ είναι ένα ε, πρόβλημα, δεν μας εκπλήσει με βάση και τα περσινά προβλήματα. Έχουμε και το περσινό μας ψήφισμα και θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην Ευρωπόλ. Δηλαδή η ΣΕΠΟΛ έχει λόγο ύπαρξης ως εξωτερικός, ως ανεξάρτητος οργανισμός, δεν μπορεί να τον απορροφήσει η Ευρωπόλ. Μπορείτε να μου απαντήσετε παρακαλώ πολύ σε αυτό. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Σταυρακάκη για τον οργανισμό φαρμάκων. Επαναλαμβάνω και τη δική του ερώτηση για την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ε, το έδαφος είναι πάρα πολύ ολιστήρο και ευαίσθητο και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι 100% ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί είναι ακέραιες και ανεξάρτητες. Και θα ήθελα παρακαλώ και σε αυτό μια απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρακάκη θα ήθελα να πω το εξή. Το τελευταίο διάστημα ε, ο κύριος Σταυρακάκης μίλησε για την ΕΜΕΑ και για την ΕΦΣΑ, για τον Οργανισμό Φαρμάκων και τον Οργανισμό ε, Ασφάλειας Τροφίμων ως προς την ανεξαρτησία των ε, εμπειρογνωμών. Για την ΕΦΣΑ, για την ασφάλεια τροφίμων, η αιτία σε αυτή κατηγορία, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι τόσο βάσιμη όσο στην ΕΜΕΑ. Στην ΕΦΣΑ ποιο ήταν το θέμα. Αυτοί που συμμετείχαν στο Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπούν συμφέροντα. Μα αυτή την επιτροπή τη λένε επιτροπή των stakeholders, των ενδιαφερομένων. Στην ΕΜΕΑ, στον Οργανισμό Φαρμάκων, είναι διαφορετική κατάσταση. Ήταν ε, ε, ανεξάρτητη σε αυτή που έπρεπε να βρούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά τέτοιοι και φτάνουν εκεί εκπρόσωποι εταιριών και επηρεάζουν πάρα πολύ τα πράγματα της αδειοδότησης φαρμάκων. Γενικά λοιπόν έχουμε μεγάλο έλλειμμα σε όλους αυτούς τους οργανισμούς ε, ως προς την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων και των μελών που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια, εποπτικά συμβούλια και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει πιο σαφείς κανόνες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Τόμας τον εκτιμώ πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, ε, της ΕΜΕΑ, ε, δέκα χρόνια έστησε αυτό τον οργανισμό και είναι πραγματικά άψογος, δεν ε, έχει κανείς να του προσάψει τίποτα χωρίς όμως κανένα χρόνο ε, κανένα διάστημα έτσι cooling off να αφήσει λίγο χρόνο να περάσει για να λάβει νέα ευθύνη και νέο αξίωμα πήγε κάπου αλλού αμέσως δεν υπήρχε λοιπόν ε, κανόνας αυτό τον οργανισμό. Ε, όπως ισχύει για τους επιτρόπους, ξέρετε, έχουν ένα κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο συζητούμε τώρα ε, για να τον αναδιαμορφώσουμε και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχουν τέτοιοι κανόνες γιατί δεν υπάρχουν για τους οργανισμούς. Γι' αυτό και η έκθεση του συναδέλφου Σταυρακάκη είναι ιδεώδης βάση έτσι ώστε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ακριβώς αυτό, να ελέγξει όλους τους κανόνες που ισχύουν, ε, όλους τους εκπροσώπους συμφερόντων ακριβώς και προσεκτικά και στην περίπτωση που ε, έχουμε ασυμβίβαστο να ε, αναλάβει και τη δέουσα δράση. Ευχαριστώ πολύ. Μακοβέη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμμερίζομαι την άποψη των συναδέλφων στην αξιολόγηση και στα αιτήματα σχετικά με την απαλλαγή των οργανισμών. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικό να συζητήσουμε σε σχέση με όλους τους οργανισμούς. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική διαφάνεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ε, στον ιστότοπο οι προϋπολογισμοί τους, όλες οι δραστηριότητες, ε, τα έσοδα, τα έξοδα. Για το προσωπικό το πρέπει να υπάρχει περιτροπή του προσωπικού από έναν οργανισμό στον άλλον ή σε άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον ιδιωτικό τομέα, στον ίδιο τομέα δραστηριοτήτων. Πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες. Ζήτησα από την Επιτροπή αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με τους οργανισμούς, αλλά δεν έλαβα ε, απάντηση. Αλλά δεν πρέπει να είναι εμπιστευτικέ αυτές οι ε, πληροφορίες ως θέμα αρχής. Ε, δεν είναι προστασία δεδομένων αν έχουμε τα ονόματα ατόμων που εργάζονται σε δημόσια όργανα. Υπάρχει και το γενικό θέμα σχετικά με την διαχείριση, την δίκηση των οργανισμών. Θα πρέπει να ε, σκεφτούμε ίσως ένα κοινό διοικητικό συμβούλιο. Έχουμε διοικητικό συμβούλιο για κάθε οργανισμό, σε κάθε διοικητικό συμβούλιο έχουμε εκπροσώπους των 27 κρατών μελών και καμιά φορά ε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ε, πολυπληθέστερο, έχει πιο πολλά μέλη από τα μέλη του προσωπικού που εργάζεται στον οργανισμό. Καλύτερα να έχουμε ένα κοινό Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερες, περισσότερους οργανισμούς των οποίων το θέμα είναι σχετικό, παραμπτός χάρη στον τομέα, τον δικαστικό. Θα πρέπει επίσης να έχουμε συντονισμό, καλύτερο προγραμματισμό και πάλι συντονισμό των δραστηριοτήτων σε έναν δεδομένο τομέα. Επίσης, σε σχέση με την ΣΥΠΟΛ, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Δεν θα επαναλάβω τα όσα συζητήσαμε. Συμφωνώ πλήρως με την αναβολή της απαλλαγής, αλλά θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι το 2007 η μεταφορά ήταν 41,5%, το 2008 31%, το 2009 33%. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, για ένα ε, ψηλό ποσοστό μεταφορών για πολλές περιόδους. Για μένα λοιπόν το θέμα αυτό δεν ξέρω αν θα, θα αυξηθεί η χρηματοδότηση ή θα πρέπει η χρηματοδότηση να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Θα ήθελα επίσης, και αυτή είναι το τελευταίο μου σημείο, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της συγχώνευσης της, ε, της CIPOL με την Europol, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας με την Europol. Αυτό το θέμα έχει ήδη αναφερθεί. Η Κομισιό έδωσε ευνοϊκή απάντηση, αλλά απορρίφθηκε από το Συμβούλιο, από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα αυτό να συζητηθεί ε, και μερικές από τις τροπολογίες μου αναφέρονται σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία και η Ευρωπόλ έχουν συμπληρωματικές δραστηριότητες και η ιδέα ε, είναι να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία στην Ευρωπόλ. Αυτό θα μειώσει τα, τις δαπάνες και θα ε, δώσει ε, προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση των των αξιωματούχων της Ευρωπόλ. Ποιος κάνει την εργασία, την διοκτική δραστηριότητα και ποιο δίνει συμβουλέ σχετικά με την εκπαίδευση. Ε, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση για τη ΛΥΜΠΕ. Εδώ συζητούμε για τα δημοσιονομικά θέματα, αλλά έχουν άμεση σχέση και τα δύο θέματα μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Σταυρακάκη για την πολύ καλή εργασία που επετέλεσε για αυτήν την απαλλαγή των οργανισμών. Είναι σημαντική εργασία, κάτι ξέρω από αυτό. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την συμβολή του στην εργασία της Επιτροπής μας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Δύο μικρές παρατηρήσεις που είναι όμως δευτερεύουσες. Θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες δευτερεύουσας σημασίας. Δεν θα ήθελα η απαλλαγή 2009 για να ε, συγχαρούμε τον νέο διευθυντή για τα όσα έχει κάνει σχετικά με την εργασία το 2010. Ε, προτείνω να βάλουμε μερικές ε, τροπολογίες στις, στα ε, συγχαρητήρια του Διευθυντή για την εργασία του 2009 και κάτι που λείπει βρίσκω ότι είναι εκτός τόπου η παράγραφος 19 χαίρεται για την πρωτοβουλία της Ακαδημίας ε, να παρέχει ε, την τελική έκθεση αξιολόγησης ε, για την απαλλαγή που κάπως δίνει διδάγματα για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Να δίνει, να, να δίνει μαθήματα διαφάνεια στους άλλους οργανισμούς η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Αυτό μου φαίνεται λίγο εκτός τόπου λόγω της ε, συμπεριφοράς της Ακαδημίας το 2007, 2008 και 2009. Αλλά ε, είναι δευτερεύουσα σημασία αυτές οι παρατηρήσεις. Ε, το θέμα του οργανισμού φαρμάκων είναι σημαντικό. Τι συνέβη βεβαίως σε σχέση με την απαλλαγή την περσινή, το ελεγκτικό συνέδριο δεν ανέφερε τη σύγκρουση συμφερόντων που υπήρχε με ορισμένα μέλη του προσωπικού και εμπειρογνώμονες. Το ανακαλύψαμε φέτος με την έκθεση ε, του, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου και έχετε δίκιο ε, που αναφέρεται ότι δεν έχουμε για όλους τους οργανισμούς την έκθεση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου θα πρέπει πριν από κάθε απαλλαγή να έχουν αυτές τις εκθέσεις, γιατί έχουμε μόνο την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι όλο και πιο ε, περιορισμένη από χρόνο σε χρόνο, ενώ οι εκθέσεις που έχουμε τυχαία, είχαμε αυτή την έκθεση σε σχέση με τον οργανισμό φαρμάκων, μας παρέχουν πάρα πολλές πληροφορίες και χάρη σε αυτή την έκθεση και ευχαριστώ την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου που μας έστειλε μέσω ενός διάβλου κάπως περίεργου, αλλά αντιληφθήκαμε φέτος ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διαφάνειας με ορισμένους εμπειρογνώμενες και μέλη του Οργανισμού Φαρμάκων. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει ε, μια ιδιαίτερη βαθμολογία ως προς την εφαρμογή των κανόνων του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, ε, ότι υπάρχει ανεντιμότητα αλλά τι διαπιστώνουμε εδώ, διαπιστώνουμε ότι η ανθρώπινη υγεία είναι το ζητούμενο πολύ περισσότερο από την ανεντιμότητα ε, και έχουμε στην Γαλλία μια υπόθεση που ίσως μερικοί διάβασαν στα εφημερίδες, την υπόθεση του Mediator που και το αναγνώρισε το εργαστήριο χτες το βράδυ στην Εθνοσυνέλευση εφόσον υπάρχει, έχει αρχίσει η προσφυγή αναγνωρίστηκε ότι υπήρχαν 38 θάνατοι λόγω του φαρμάκου Μεντιατόρ που το Ben είναι το, το όνομα του γενοσύμου ε, και ορισμένα άτομα είχαν ζητήσει το 98 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μια έρευνα η έρευνα αυτή άρχισε, δύο εμπειρογνώμενες του Οργανισμού Φαρμάκων είχαν ασχοληθεί με την έρευνα αυτή, ένας Ιταλός και ένας Γάλλος και ε, δεν υπήρξε και δεν έγινε καμία προσφυγή μετά την έρευνα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εγώ διαρωτώ με σε τι χρησιμεύει αυτή, ο οργανισμός, πού είναι η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων του προσωπικού, υπάρχει σύγκρουση συμφορώντων, το πρόγραμμα παραμένει, το πρόβλημα παραμένει ε, στην Γαλλία ε, το, σε ορισμένα κράτη-μέλη βαθμία αυτό το φάρμακο, αλλά ε, τι έγινε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων, από ό,τι ξέρουμε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, δεν τηρήθηκαν μέσα στον οργανισμό αυτό. Βεβαίω, συμφωνώ πλήρω με εσά, κύριε Σταυρακάκη, για να αναβάλουμε την απαλλαγή. Ακόμη και να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και εγώ σας προτείνω να έχουμε μια ακρόαση στην Επιτροπή μας με τον Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι όπως και πέρσι το είχα πει για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, συνήθως ε, καταλογίζουμε τα πάντα ε, στο Διευθυντή, ενώ υπάρχει μια μεγάλη χαλαρότητα και επίοικια ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα ήθελα να έχουμε μια ακρόαση στην Επιτροπή μας. Σας το προτείνω, σας το ζητώ εξάλλου. Ευχαριστώ, συνάδελφος Τσέσκοβα. Ευχαριστώ πολύ. Έλαβα τον λόγο αρκετά αργά και πάρα πολλοί προλαλήσαντες ε, ήδη ανέφεραν τα όσα ήθελα εγώ ίδια να πω, αλλά θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό ε, κοινών επιχειρήσεων, κοινών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ από τότε που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κατάσταση σχετικά με τον αριθμό των οργανισμών και τη λειτουργία τους είναι πάρα πολύ υψηλός. Και νομίζω ότι για τον Ευρωπαίο πολίτη Όλη αυτή η δομή δεν είναι διαφανής. Και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε πράγματι να κάνουμε την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών και να διαρωτηθούμε οι δραστηριότητες τους είναι πραγματικά απαραίτητες. Δεν μπορεί να υπάρξει συγχώνευση ανάμεσα σε ορισμένους οργανισμούς και πιστεύω ότι πράγματι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ίσως δεν αφορά την συζήτηση που έχουμε για την απαλλαγή το θέμα αυτό, αλλά είμαι πεπισμένη ότι πρόκειται, ότι είναι ένα θέμα συζήτησης σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια συζήτηση και νομίζω ότι ορισμένοι προλαλήσαντες το ανέφεραν το θέμα το δικαίως. Σας προτείνω λοιπόν να ε, βάλουμε σε αυτήν την έκθεση μια προσθήκη και να πούμε ότι ίσως θα έπρεπε ο όχι να αυξάνεται ο αριθμός των οργανισμών, αλλά να εξορθολογήσουμε τον αριθμό αυτών των οργανισμών και τη λειτουργία του. Σας ευχαριστώ. Ε, ähm, κύριε Γκάιερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο του Σταυρακάκη για την πολύ καλή δουλειά του και να υπογραμμίσω ότι συμμερίζομαι τις προτάσεις του και τα όσα είπε. Ανισχώ όμω για ένα συγκεκριμένα. Είναι ένα είδος ομοιομορφίας για όλους τους οργανισμούς όταν συζητάμε εδώ στην Επιτροπή μας. Υπάρχει λόγος που ιδρύσαμε τους οργανισμούς αυτούς και τον καθένα ξεχωριστά. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι όλα τέλεια και θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αλλά η συζήτηση που ανάγεται και να περιορίζεται στο γεγονό ότι έχουμε υπερβολικό αριθμό οργανισμών χωρί συγκεκριμένα επιχειρήματα για να τεκμηριωθεί αυτό, για να στοιχειοθετεί ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί που περιτεύουν και τι θα γίνει με το αντικείμενο τη δουλειά στο μέλλον, πού θα το πάμε. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση με τρόπο επαρκή για μένα. Γι' αυτό και η σοβαρότητα της αντιμετώπισης ε, της Επιτροπής μας των οργανισμών αυτών θα αυξηθεί μόνο εφόσον με συγκεκριμένα στοιχεία και του ελεκτικού συνεδρίου και των εσωτερικών ελεκτών τεκμηριώσουμε ε, την κατάσταση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε όποτε θέλετε συζήτηση γενικά ποιοι οργανισμοί πληρούν το έργο τους, το καθήκον τους και ποιοι όχι, ποιοι πρέπει να καταργηθούν κτλ. Αλλά να γίνουν αυτά με στοιχεία, με γεγονότα, όχι μόνο σε αυτή εδώ την Επιτροπή και στις ε, επιμέρους αρμόδιες και υπό το φως των ειδικών εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Και θα έρθει και φέτος η ειδική έκθεση συγκεκριμένη. Αυτά τα είπα περίπου ακριβώς τα ίδια και την περασμένη φορά που συζητούσαμε για τους οργανισμούς. Και σχεδόν αντανακλαστικά γίνεται η συζήτηση πλέον. Ότι η πρώτη διαπίστωση βγαίνουν και λένε ορισμένοι ότι είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός και δεύτερο να τα ελέγξουμε λέτε ή λένε ορισμένοι. Όχι, εγώ το λέω αντίστροφα. Πρώτα να ελέγξουμε και μετά να καταλήξουμε εάν είναι υπερβολικά πολλοί και περιτεύουν κάποιοι οργανισμοί. Έτσι, με την αντίστροφη σειρά. Και μετά να καθορίσουμε ξεκάθαρα και τι ευθύνε και τι αρμοδιότητε. Και να μην απαλλάσσονται τα κράτη-μέλη από τι ευθύνε του. Αν δούμε το πρόβλημα στην αστυνομική ακαδημία δεν είναι καινούριο στη ΣΕΠΟΛ. Αυτό διονύζεται, συνεχίζεται και δεν έχει λυθεί εντελώ ακόμα. Γιατί αυτό, διότι ε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτείται από εκπροσώπους 27 κρατών μελών και απέτυχε εκτρά. Και δεν ενθουσιάζονται τα πλήθη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια, παρά μόνο τη στιγμή που παίρνει την έδρα η χώρα τους, ξεσπάει τρομερός λαϊκός ενθουσιασμός και μετά τον ξεχνάνε τον οργανισμό. Ποιος φέρει την ευθύνη για την παρατήρηση και την παρακολούθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της λειτουργίας των οργανισμών αυτών. Ευχαριστώ. Ο Σάφος Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία πράγματα, λίγα μόνο. Έχουν υποθεί πολλά και με έχουν καλύψει και πολλά και συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σταυρακάκη, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση του και τον στηρίζει και η ομάδα μας και τις συστάσεις του. Σε δεύτερο λόγο να περάσω στις παρατηρήσεις που έκανε και η κυρία Ματιού. Αυτά που είπε δηλαδή ότι ε, ισχύουν, είναι ε, πολύ σωστά και να το κοιτάξουμε στους συντονιστές, κύριε Πρόεδρε, μαζί με τον εισηγητή, σε περίπτωση ε, που αναβάλουμε την απαλλαγή ή δεν τη δώσουμε για τον οργανισμό φαρμάκων, να το συζητήσουμε πολύ καλά να συνεννοηθούμε με τον ε, εισηγητή ή συντονιστές η ακρόαση μου φαίνεται μία από τις τεχνικές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει το θέμα και μεθοδικά και παρακαλώ να το δούμε και συμφωνώ και υποστηρίζω την κυρία Ματιό. Και ένα τρίτο, συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε μόλις ο κύριος Γκάιερ. Να κοιτάξουμε πώς ε, θα γίνει ευρύτερη συζήτηση ε, από τη στιγμή που θα έχουμε δώσει τη μία απαλλαγή μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσουμε να συζητάμε για την επόμενη. Ε, να κοιτάξουμε το ρόλο των οργανισμών. Είναι καλοί όλοι οι οργανισμοί, κάνουν τη δουλειά τους, μπορούν ορισμένοι να συνενωθούν. Μήπως χρειάζεται να τους ξαναεξετάσουμε. Μια πολύ εκτενή συζήτηση, αλλά ξεχωριστή. Αυτό δεν είναι αντικείμενο της απαλλαγής, ανάμεσα στις δύο συζητήσεις, αυτής της απαλλαγής και της επόμενης. Ας ακούσουμε και τους, ε, τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Οσία. Έχετε το λόγο. Αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, είναι τιμή μου, τιμή του Ελεγκτικού Συνέδριου να παρίσταται στην αίθουσα για να απαντήσει σε ερωτήσει που έθεσαν ο συγητής κύριος Σταυρακάκης και η συναδελφή του μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Σταυρακάκη για το έργο του, για τόσες πολλές εκθέσεις απαλλαγής. Είχαμε καλή συνεργασία με τον κύριο Σταυρακάκη, με τον βοηθό του κύριο Λατούδη και με την δίκηση, ιδιαίτερα την κυρία Μενάλτη και την ομάδα της. Πριν από εννέα μήνε έγινα μέλο του Ελεκτικού Συνέδριο υπεύθυνο για, τα, για τις υπηρεσίες τον Ιούλιο. Άρχισα να ε, α, α, α, αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον τη επιτροπή σα για την λειτουργία των υπηρεσιών και μπορεί να ενισχυθεί το έργο των υπηρεσιών, να βελτιωθεί προκειμένου τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε αυτές να πιάνουν τόπο για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο ο οποίος εμπιστεύεται τα χρήματά του στην Ένωση να τα διαχειριστεί σωστά για λογαριασμό του. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που έθεσε ο κύριος Σταυρακάκη σε σχέση με την απαλλαγή. Καταρχήν ήθελα να σας θυμίσω ότι το 2008, στην απαλλαγή του 8 μάλλον, μας ζητήσατε το Κοινοβούλιο να μελετήσουμε ορισμένους δείκτες αποδοτικότητας σε σχέση με τους οργανισμούς και πολύ πρόσφατα, πριν από δύο μήνες το Δεκέμβριο, η Επιτροπή ζήτησε από το Ελεκτικό Συνέδριο να κάνει μια ανασκόπηση της δαπάνης των οργανισμών. Έχουμε την ειδική έκθεση Cost Benchmarking στις, ε, στους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρεται στην έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη. Και χαίρομαι για το ότι μπορώ να σας πω ότι η δουλειά έχει αρχίσει, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και θα το δημοσιεύσουμε το φθινόπωρο. Με ικανοποίηση παρακολούθησα μια συνάντηση των εκπροσώπων των αντιπροσωπιών των Εθνικών Κοινοβουλίων στην θεσμική ομάδα χθες όπου αναφέρθηκε το εύρος της εργασίας αυτής και το χρονοδιάγραμμα. Το αίτημα προς το ηλεκτρικό συνέδριο και η απάντησή μας είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπω σας είπα, για να πιάνουν τόπο τα λεφτά του φορολογούμενου. στην διαχείριση των οργανισμών. Η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών έκανε δύο προτάσεις. Πρώτον, στο μία ε, ανασκόπηση της ε, περιπτώσης σύγκρουσης συμφερόντων, απαντήσαμε υπεύθυνοι, ως υπεύθυνο για τα ε, ρυθμιστικούς οργανισμούς ε, είμαι αρμόδιος να μελετήσω ακριβώς αυτό το έργο, τι κατεύθυνση θα πάρει και θα το συζητήσω καταρχήν με τους αδέρφους μου στο ελεγκτικό συνέδριο με πνεύμα συνεργασίας. Ακόμα δεν έχουμε μπει μέσα στο, σε βάθος σε αυτή τη δουλειά προκειμένου να ε, συνεργαστώ με τους αδέρφους. Επαναλαμβάνω το πνεύμα θα είναι πνεύμα θετικό με βάση το αίτημά σας ε, σχετικά με την εργασία πέρυσι. Ο κύριος Σταυρακάκης έθεσε μια ερώτηση σχετικά με την υπηρεσία για την Ευρατόμ. Η Ευρατόμ είναι ένα σημαντικός οργανισμός, ελέγχει την παραγωγή, την παροχή και τη μεταφορά ουρανίου και προϊόντων ουρανίου. Είναι ένας παλιός οργανισμός δεν έγινε με νομοθέτημα όπως άλλοι οργανισμοί. Το δημιούργησε η ίδια η συνθήκη. Είναι ένα ειδικού τύπου οργανισμός. Η Επιτροπή το ελέγχει. Η Επιτροπή μπορεί να βγάλει οδηγίες, μπορεί να προβάλλει βέτο στις αποφάσεις του οργανισμού, ορίζει το προσωπικό, πληρώνει το προσωπικό. Αλλά τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός αυτός δεν είχε προπολογισμό. Όλες οι δαπάνες σχετικές με αυτόν γίνονται από την Κομισιόν για λογαριασμό του οργανισμού. Είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση κύριε Πρόεδρε. Οι λογαριασμοί είναι παγωμένοι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προπολογισμό για τον οργανισμό από το 2007 και μετά. Άρα ο, ο, οι λογαριασμοί είναι απλοί, γιατί πολύ λίγε πράξει περνάνε μέσα από του λογαριασμού αυτού, γιατί δεν υπάρχει προπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί είναι ε, νόμιμοι, ε, κανονικοί, υπάρχει η κοινωτική νομοθεσία ε, όσον αφορά όρους χρημάτων, το ποσό είναι μικρά. 200.000 ευρώ περίπου σε, για διοικητικές δαπάνες που επαναλαμβάνει το, το διαχειρίζεται η Κομισιόν. Το καθεστώς ε, του οργανισμού λέει ότι αυτέ τι 200.000 θα πρέπει να του δαπανά ο οργανισμός και όχι η Κομισιόν. Στο ηλεκτρικό συνέδριο το συζητήσαμε το θέμα αυτό με τον οργανισμό και προτείναμε λύση με αλλαγέ στο καταστατικό ο διευθυντής του οργανισμού είναι σε θέση σήμερα να σας ε, ε, πληροφορήσει πώς έχουν τα πράγματα. Πρόκειται για μικρές αλλαγές με βάση τη νομική συμβουλή που πήραμε. Συμπληρωμα... Ε, ε, η σχέση για την Ευρωτόμ είναι νόμιμη κανονισμή. Το, τα ποσά σε χρήμα είναι μικρά. Όπω είπε και ο κύριος Σταυρακάκη στην έκθεσή του, η κατάσταση ωστόσο θα πρέπει να ε, γίνει πιο ομαλή, πιο κανονική και το τονίζουμε αυτό στην έκθεσή μας. Η άρεστη συμβολή με εικόνα από τους ε, συναδέλφους σας στην Επιτροπή, ήθελα να επισημάνω, κάνουμε, θα κάνουμε μια έκθεση με δείκτες σχετικά με το κόστος, cost benchmarking, και έτσι θα καλύψουμε κάμπος από τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι συνάδελφοί σας σε σχέση με την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση όσον αφορά τους οργανισμούς. Αυτό αφορά τη διακυβέρνηση, governance, και τις δαπάνες. αυτό που πρότεινε η Επιτροπή σας η εργασία σχετικά με την σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης σχετικά με την περίοδο που χρειάζεται για να ε, καλυφθούν τα δύο κενά, αυτό που λέμε cooling off period». Η μελέτη για τους δείκτες σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Γκίρ ε, και σε σχέση με τη συμφωνία για την SIT ε, Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν τυχόν έχετε ερωτήσεις αυτή τη στιγμή για τους ε, ε, διάφορους οργανισμούς. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Πρόεδρος, ο κύριος Νόακ τώρα και αυτός από το ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θίξω και εγώ μερικά θέματα. Όπως ξέρετε έχουμε μια μοιρασμένη ευθύνη μεταξύ των υπηρεσιών και των κοινών των joint undertakings όπως τα λέμε από την σύνθεση τους και το στόχος τους είναι ένα διαφορετικό ε, όργανο και δεν μπορούν να συγκριθούν με τους οργανισμούς, τα agencies. Τα τελευταία τρία χρόνια υπεύθυνο για τον έλεγχο αυτών των ε, κοινοπραξιών, joint undertakings, την επόμενη χρονιά ο κύριος Μπάλκο, ο οποίος είναι δεύτερος από τα αριστερά μου, θα είναι ο αρμόδιος στο ελεκτικό συνέδριο για τις ε, κοινοπραξίες, joint undertakings. θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κύριος ε, Σταυρακάκης μας έδωσε μια άριστη βάση για συζήτηση και αποφάσεις σε σχέση με, τις, με την απαλλαγή των ε, κοινοπραξιών με βάση τις δικές μας ε, εκθέσεις ελέγχου. Ένα μόνο θέμα θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Σταυρακάκη. Μίλησε για τις δυσκολίες που συνήθως υπάρχουν στην αρχή που έχει μια εταιρεία με κοινοπραξία. Στις δικές μας εκθέσεις εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας αλφα βαθμός μειωμένη δαπάνη στην αρχή στην εκτέλεση του προπολογισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τι πιστώσει πληρωμών. Αυτή η μειωμένη δαπάνη στην αρχή δικαιολογείται λόγω της πολιετούς φύσης των προγραμμάτων και από την καθυσέρηση στην εκτέλεση των διαφόρων έργων. Αυτό το ποσοστό αυτός, που εμφανίζεται στην αρχή λειτουργίας υπό δαπάνης, το πούμε, του προπολογισμού, χαρακτηρίζει τις περισσότερες κοινοπραξίες που ξεκίνησαν τη δραστηριότητα του 2009. Τι σημαίνει αυτό. Όσο θα αυξάνεται η εμπειρία από το έργο, από την διαχείριση των στόχων, τα προβλήματα αυτά ευελπιστούμε ότι θα μειώνονται σε μεγάλο βαθμό. όσον αφορά προβλήματα ε, παρατυπίας ημί. Σε μερικές περιπτώσεις οι γενοπραξίες, ως απαιτείται δεν έχουν την ίδια ρύθμιση προσανατολισμένη παράλληλα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης. Τα προβλήματα όμως και αυτά με το χρόνο μειώνονται. Πριν από λίγο διάβασα ένα κείμενο έγκριση για την ε, κοινοπραξία Clean Sky θα έχει το δικό της κανονισμό όπως ε, πρότεινε ο κύριος Μπάλκο και όπως επιβάλλεται και επαναλαμβάνουμε ότι τον τρόπο αυτό τα προβλήματα θα μειώνονται και είναι στο σωστό δρόμο οι κοινοπραξίες αυτές. Ευχαριστώ. Ο Διευθυντής της Ευρατόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η παρουσίαση που έγινε από τα δύο μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου με βρίσκουν τελείως σύμφωνο με την έννοια ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη είτε η ε, πραγμα τικότητα να συνάδει με το καταστατικό ή το καταστατικό με την πραγματικότητα. Θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρίας αυτής, διότι σχετικά με τον οργανισμό αυτό βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Εάν πάρουμε τον στόχο που είναι να φροντίζει για τον εφαδιασμό όλων των χρηστών πυρηνικών υλικών και να μην υπάρχει διάκριση. Η μη διάκριση είναι βεβαίως ε, σημαντικό. Είδατε τις ε, ατέρμονες ε, συζητήσεις για το αέριο, για το πετρέλαιο, για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Το τρίτο πακέτο ενέργειας θα έλεγα ότι όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια η μη διάκριση είναι μία από τις βασικές ευθύνες αυτού του οργανισμού. Δεύτερο σημείο, ένα τακτικός εφοδιασμός. Τακτικός σημαίνει ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Το να συζητούμε σήμερα για ασφάλεια είναι κάτι το εξ, πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι όσον αφορά στον πυρηνικό τομέα, εγγυόμεθα 30% του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό. Θα έπρεπε λοιπόν να συμφωνήσετε ότι για 200.000 ευρώ κατέτος το να έχει κανείς μια τέτοια ευθύνη μας κάνει ένα μέσο, ένα όργανο που ε, τηρεί ε, μια, τα, τις αρχές της χρηστής διαχείρισης. Ποιες είναι οι ευθύνες της, του οργανισμού. Υπογράφουμε ε, συμφωνίες εμπορικές. Έχουμε μια δραστηριότητα εμπορική. Μπορούμε ε, να έχουμε από θέματα ασφαλείας. Αν μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα για το αέριο και το πετρέλαιο, δεν θα βρισκόμαστε στην κατάσταση που έχουμε σήμερα για τους δύο αυτούς τομείς έχουμε σημαντικές συζητήσεις. Έχουμε ένα συμβουλευτικό συμβούλιο με εκπροσώπους των κρατών μέλων. Ένα μεγάλο από τους στόχους ενεργειακής πολιτικής είναι να μιλάμε με μία φωνή. Κύριε Πρόεδρε, στον πυρηνικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλο τον ε, σεβασμό ε, τον οποίον οφείλω στα κράτη-μέλη για την απόφαση του μείγματος του ενεργειακού που προβλέφθηκε στη Λισαβόνα, θα έλεγα ότι όσον αφορά τον οργανισμό διαμέσου ε, του συμβουλευτικού οργάνου μιλούμε με μία φωνή. Βλέπουμε, ε, είναι η μόνη ενεργειακή κοινοτική πολιτική που υπάρχει σήμερα ε, και που είναι η ευθύνη αυτού του οργανισμού. Η διαφάνεια προφανώς είναι σημαντικό κύριε Πρόεδρε και καταλαβαίνω πολύ καλά αυτή τη συνέλευση που το Κοινοβουλίο που ε, δίνει τόση μεγάλη ε, σημασία στους οργανισμούς και στην διαφάνεια, την τέλεια διαφάνεια του οργανισμού. Ίσως ε, να ήμασταν καθολικότεροι του Πάπα, διότι μετά τις συστάσεις ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2008 υποβάλαμε ένα ξεχωριστό δημοσιονομικό κανονισμό και δεν ξέρω αν αυτό ήταν καλό, διότι με βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε αυτόν τον κανονισμό και επιπλέον ε, ενέγραψε ε, με ένα προσυπόμνηση τον προϋπολογισμό μας. Χρειάστηκε βεβαίως να επιβιώσουμε και καταλαβαίνετε ότι εγγυόμαθα 30% του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό. Αν δεν έχουμε χρήματα δεν θα είχαμε εδώ φώτα. Νομίζω ότι από αυτήν την άποψη έχουμε προφανώς επωφεληθεί από την δημόσια γενεοδορία, μπορώ να πω, της Γενικής Διεύθυνσης Τρέν και τώρα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας με το ελεγκτικό συνέδριο μετά τις συζητήσεις που ε, είχαμε εξετάζουμε τη δυνατότητα να συνάδει η πραγματικότητα με το καταστατικό. Παρακολουθούμε με τη νομική υπηρεσία αυτήν την διαδικασία. Αν είχαμε τροποποιήσει το καταστατικό θα ε, έπρεπε να περάσουμε από το Συμβούλιο που θα είναι μια άσκηση πάρα πολύ περίπλοκη σε σχέση με τις δυσκολίες που είχαμε με το νέο καταστατικό το 2007. Αλλά τούτων λεχθέντων κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι τα κονδύλια ε, που διοχετεύονται στον οργανισμό 200.000 ευρώ σε σχέση με εκατομμύρια αν μπορούσαμε ε, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο και πετρέλαιο με 200.000 ευρώ, νομίζω ότι θα ψηφίζατε με τα δύο χέρια για μια τέτοια απόφαση. Έχουμε τον ε, Διευθυντή επίσης για την υπηρεσία τα φάρμακα. Κύριε Σταυρακάκη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που με απευθύνετε και που μετά τις 25 Ιανουαρίου έχω την ευκαιρία να σας ε, ξαναμιλήσω για τις εκθέσεις που έχουν υποβάλει ελεκτικό συνέδριο και κοινοβούλιο ε, για τον οργανισμό μας. 15 συναπτά έτη δεν γινόταν κανένας λόγος για μας ε, στην Επιτροπή σας. Γι' αυτό έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα για τη φετινή κατάσταση. Εγώ θα μιλήσω για αυτά που μας ρωτήσατε για τις προσλήψεις, μεταφορά, ε, πιστώσεων, ανάθεση, εξεγονισμών και στο τέλος ε, στη σύγκρουση συμφερόντων στον οργανισμό μας. Σωστά επικρίνεται τη διαδικασία των προσλήψεων στον οργανισμό Έχουμε βελτιώσει έκτοτε ε, τις διαδικασίες. Πολλές ε, διακόπησαν. Το προσωρινό προσωπικό, το έκτακτο, δεν έχει πρόσβαση ε, στις ευαίσθητες προφορίες. Το αποφασίσαμε ήδη από το 2009. Η βάση δεδομένων των εμπειρογνωμόνων έχει συμπληρωθεί και το 2010 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάνει τις βελτιώσεις της ε, ε, η ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα προϊόντα έχουν επίσης βελτιωθεί από το 2009 και μετά και ε, κάποιες παλινοδίες και είχατε επισημάνει το 2010 τις αυστηροποιήσαμε. Για να προστατεύσουμε τον προϋπολογισμό μας εργαζόμαστε Ε, με στερλίνες ε, και ξέρετε ότι η λία η στερλίνα και το ευρώ έχουν πολύ μεγάλες διακοιμάνσεις στην συναλλαγματική τους ισοτιμία και αυτό μας δυσκολεύει. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα σας είπα στις 25 Ιανουαρίου, να είστε βέβαιοι όμως ότι όλα τα μέτρα που προτείνει ο εισηγητής ε, και όλες οι επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες από το 2008 και ε, μετά είναι κάποια θέματα που μας έχουν απασχολήσει, δίνουμε συνέχεια και φροντίζουμε να ε, εξαλειφθούν. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά που αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, πρέπει να σας εξηγήσω κάτι ιδιαίτερα, γιατί έχει να κάνει ακριβώς με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός φαρμάκων. Κυρίες και κύριοι, όταν έρχεται μια αίτηση από μια φαρμακευτική εταιρεία σε εμά. Έχουμε 7 μήνες για να την επεξεργαστούμε ε, αυτή την αίτηση. Αυτή είναι πολύ λιγότερο από ό,τι στα κράτη-μέλη. Μέχρι και 12 χρόνια έχουμε ακούσει στο παρελθόν για τα κράτη. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο μέσα σε ένα επτάμινο να έχουμε απαντήσει. Και αν είναι ειδικέ ερωτήσεις που έχουν οι επιτροπές στις φαρμακευτικές εταιρείες σταματάμε το ρολόι και ε, κρατάει περισσότερο, 8-9 μήνες μέχρι και ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχει υποβληθεί η αίτηση και έχει επικυρωθεί, έχει κατοχυρωθεί ως έγκριση, θα πρέπει να πληρώνει η εταιρεία. Δηλαδή, από τη στιγμή που πρωτοκολλείται, ας πούμε, η αίτηση, αρχίζει να πληρώνει η εταιρεία και η εργασία. Και το 50% ε, των ε, εσόδων μας από τα τέλη αυτά πηγαίνουν στα κράτη-μέλη για να χρηματοδοτήσουμε εκεί την πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, σε αυτό το πεντάμινο, ε, ε, εισπράττουμε τέλη. Ενώ η πραγματική εργασία για την ουσία θα γίνει το επόμενο έτος. Λοιπόν, είτε θα τα εγγράψουμε αυτά στον προπολογισμό, γι' αυτό και είναι και μεγάλη μεταφορά από το ένα έτος στο άλλο. Ξέρω πώς λειτουργούμε, γι' αυτό σας λέω. Ε, τα ίδια για την αεροπορία. Πληρώνει ε, η ε, εταιρεία για να αρχίσει να εξτάζεται η αίτησή της για να κυκλοφορήσει ένας νέος τύπος αεροσκάφος στο μέλλον. Είναι μια κυλιόμενη διαδικασία που δεν βασίζεται, ούτε σέβεται αυτό το ενιάψιο που είναι ο χαρακτήρας του προπολογισμού, γι' αυτό μεταφέρεται και μετακυλείται από τον ένα στον άλλο. Για το ελεγκτικό συνέδριο είναι απαράδεκτη αυτή η μεταφορά πιστώσεων, πολύ υψηλή δηλαδή το carry-over. Αλλά αν δεν γράφουμε αυτά τα κονδύλια στον προπολογισμό, έχουμε πλεόνασμα μη απορροφηθέν, το οποίο πηγαίνει πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι μια κατάσταση lose-lose, δηλαδή και, και στις δύο περιπτώσεις είμαστε χαμένοι. Ε, και κάθε χρόνο το ζω αυτό. Και αυτό ε, πιτοπλίστων επιλέγουμε τη μεταφορά από το ένα έτος στο άλλο και ελπίζω να μας κατανοήσει το ελεγκτικό συνέδριο. Και ένα τρίτο. Αυτά για τις μεταφορές από τον ένα χρόνο στον άλλο. Ό,τι και να κάνουμε θα είμαστε χαμένοι. Μπρο γκρεμό και πίσω ρεύμα. Το τρίτο είναι οι διαδικασίε ανάθεση. Ε, έχετε δίκιο, ε, ε, κύριε Σιγητά, για τι διαδικασίε ότι υπήρξαν σφάλματα στο παρελθόν και δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να το δικαιολογεί. Βελτιώσαμε τι διαδικασίε τι κάναμε πιο αυστηρέ με ελέγχου, Ε, τώρα πρέπει να λειτουργήσουν και οι άνθρωποι αντίστοιχα. Ένα άλλο σημείο, και αυτό είναι ένα μικρό παραθυράκι τώρα στο δημοσιονομικό κανονισμό, είναι οι λεγόμενες άμεσες αναθέσεις, οι άμεσες συμβάσεις που έχουμε διαπραγματευτεί για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών ή άλλων που ήδη ισχύουν. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει αγορά ή είναι απογορευτικό το κόστος αν βγαίναμε στην αγορά και ήταν ανοιχτό ο διαγωνισμός. Αυτή η διαδικασία ε, ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος σας έχει φτιάξει ε, ας πούμε μια τράπεζα δεδομένων και η ίδια εταιρεία την παρακολουθεί κάθε χρόνο. Επί μια δεκαετία που είμαι εγώ στον οργανισμό, έχουμε διαπραγματευτεί με τις αντίστοιχες εταιρείες για ε, καλύτερες ε, προϋποθέσεις, καλύτερους όρους κλπ. Και όλα πήγαιναν καλά. Εδώ και δύο χρόνια, δεν ξέρω ποια ιδιοφυΐα το εφήβρε αυτό, κατέβασε αυτή την ιδέα, μας αναγκάζουν σε συμβάσεις που διαπραγματευόμαστε άμεσα να ε, ε, επιβάλλουμε την ίδια διαδικασία. Εγώ δεν θέλω να επικρίνω το δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά είναι και δική σας αρμοδιότητα να βελτιώσετε το δημοσιονομικό κανονισμό και αν μου επιτρέπετε να το πω. Σε περίπτωση που διαπραγματευθήκαμε άμεσα μία σύμβαση σε αυτή ε, την υπόθεση, πρέπει να πάμε στην εταιρεία και να της πούμε. Βάλε το αποτέλεσμα σε δύο σφραγισμένους φακέλους, στείλτο, στην εταιρεία, στον οργανισμό να βάλουμε και προθεσμία πότε θα ανοιχτούν οι σφραγισμένοι φάκελοι, που βεβαίως δεν έχουμε γνώση αυτών, πότε θα ανοιχτούν οι φάκελοι σε κάποια επιτροπή και μετά να ορίσουμε και ελεγκτική επιτροπή να τη συστήνουμε γι' αυτό για να αξιολογήσει ξανά τα γνωστά κατά τα άλλα αποτελέσματα του διαγωνισμού και μετά να κάνουμε και διαδικασία επιλογής για μια επιλογή που δεν υφίσταται αφού ένας είναι ο συμβαλόμενος εδώ και χρόνια. Κυρίες και κύριοι, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και ε, λιγότερο γραφειοκρατικοί, αλλά τώρα μας υποχρεώνουν σε τέτοιες καταστάσεις τύπου Κάφκα. Τι να κάνουμε κι εμείς, παρακαλώ, κοιτάξτε εσείς αυτό το πρόβλημα και διορθώστε το. Και ένα τελευταίο για τον κώδικα συμπεριφοράς και τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο οργανισμός, πολύ περισσότερο ίσως από κάποιου άλλους οργανισμού, ε, καλείται ιδιαίτερα να προλαμβάνει και να αποφεύγει ε, συγκρούσεις συμφερόντων και στο προσωπικό της και σε εμπειρογνώμονες αλλά και σε εθνικούς εμπειρογνώμονες που δουλεύουν στις χώρες τους, είναι αποσπασμένοι αλλά δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους στον οργανισμό. Και αυτό ισχύει και για τους πρώην υπαλλήλου. Πρέπει να σας πω ότι ανέκαθεν υπήρχε κώδικα συμπεριφοράς και δεντολογίας και πολιτική ε, ή ε, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στον οργανισμό μας. Διαπιστώθηκαν κατά καιρού παραβιάσεις στο παρελθόν. Αυτό δεν ήταν ει βάρο το οργανισμό αυτού καθ' αυτού, αλλά παραβιάσεις έχουν διαπιστωθεί. Αυτός ο κώδικας συμπεριφορά, αυτή η δήλωση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, βασίζεται σε εθελούσια δήλωση του ενδιαφερομένου παντού, σε άλλου του οργανισμού. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος κάθε φορά να δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο, καμία σύγκρουση συμφέροντο. Εμεί αστυνομία δεν έχουμε. Ούτε υπηρεσίε ασφαλεία που κάθε φορά να ελέγχει τα όσα έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενο. Και κατά τα άλλα δεν προβλέπεται αυτό, δεν είναι δουλειά μα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, χρειαζόμαστε πολιτική καθοδήγηση τι θα κάνουμε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση 27 κράτη-μέλη. Πώς να ελέγχεις το υπόβαθρο, το background του κάθε εμπειρογνώμονα σε περίπτωση που μας ζητηθεί και δεν συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στην αρχή της εμπιστοσύνης. Και προς το παρόν, το είπε και πολύ σωστά ο εισηγητής, προς το παρόν οι κανόνες αυτή, της απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων ενισχύονται, οξύνονται. Αλλά να σας πω το εξή ξεκάθαρα το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δεχτεί αυτούς τους όρους και να τους εγκρίνει. Και δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη στο Διοικητικό μας Συμβούλιο να ενταθούν και να ενισχυθούν αυτές οι ρυθμίσεις με αυτή την αυστηρότητα. Για ποιο λόγο. Γιατί σε, υπάρχουν χώρες ε, όπου υπάρχει αυτή η κουλτούρα, η πολιτική επιθυμία να συνεργάζεται η βιομηχανία με την πολιτική. Υπάρχουν χώρες που είναι και υπερήφανοι ε, που συνεργάζονται οι πολιτικοί με τους επιστήμονες και με τη βιομηχανία. Και όταν τους συζητάμε μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας ω ανεξάρτητοι. μα λένε βεβαίω, αλλά έχω κάνει πριν από χρόνια για την ΑΒΓ εταιρεία ε, αυτή την γνωμοδότηση. Είναι ζυξάκ αυτό το πράγμα, δεν είναι άσπρο μαύρο. Ε, αλλά ενισχύσαμε, κάναμε πιο αυστηρούς τους κανόνες και τους κρίναμε και για το προσωπικό μας και για τον οποιοδήποτε πατάει το πόδι του στον οργανισμό. Ένα τελευταίο. Τώρα. Για το Μετιατόρ. Βεβαίω, υπέστη κριτική και ο οργανισμός μας και σε σχέση με τη σύγκρουση φερόνων, Αλλά κυρία Ματιού, Μπορώ να σας διαβεβαίωσω, ο οργανισμός σεβάστηκε όλους τους κανόνες και τους στήρισε όλους τους υφιστάμενους κανόνες. Δυστυχώς το προϊόν είναι εθνικό σε κυκλοφορία, σε αγορά της χώρας. 90% των φαρμάκων στην Ευρώπη κυκλοφορούν ε, σε επίπεδο κράτους, μέλους και μόνο το 10% χρειάζονται πανευρωπαϊκή αδειοδότηση γιατί αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο τα τελευταία 15 χρόνια. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Τα πρώτα χρόνια ήμασταν στριμωγμένοι στον τοίχο. Είχαμε 46 πάρα πολύ υπερήφανους, ε, ανεξάρτητους εθνικούς ε, οργανισμούς φαρμάκων που ε, γινόντουσαν έξαλλοι κάθε φορά που θεωρούσαν ότι μπαίναμε στα χωράφια τους και μας φέρναν την αρχή της επικουρικότητας απέναντι. Δηλαδή κάντε την ευρωπαϊκή σας δουλειά και αφήστε μας μόνους μας στις χώρες μας να κοιτάμε τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά μας και μην ανακατεύεστε. Το, 80, το 98 και το 99 αυτή ήταν μια άποψη που κυκλοφορούσε πολύ ευρύτερα και η ΕΜΕΑ δεν είχε δυνατότητα καν, άσε που δεν είχε κανένα δικαίωμα, δεν είχε καν τη δυνατότητα να μπαίνει σε ζητήματα παρακολούθησης φαρμάκων που κυκλοφορούσαν στις αγορές των κρατών μελών. Και ένα τελευταίο. Πώς εφαρμόζουμε τον κώδικα διοντολογίας και συμπεριφοράς σε αφορά τα μέλη του προσωπικού μας, υπαλλήλου δηλαδή, που συνταξιοδοτούνται ή φεύγουν από την, ε, τον οργανισμό. Ε, σωστά υπόθηκε ότι είναι πάρα πολύ θολή η νομική βάση και ασαφής. Ωστόσο, στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων μας υπάρχει το άρθρο 16, το άρθρο 16 που υποχρεώνει το πρώην προσωπικό να σέβεται ε, τον κώδικα συμπεριφοράς και να ενημερώνει τον οργανισμό για τις νέες δραστηριότητες που ε, αναλαμβάνει. Αυτό συνέβη πρώτα με πολύ γενικό τρόπο και στη συνέχεια με πολύ ειδικό και συγκεκριμένο. Και επειδή συνέβη σε ειδικό και συγκεκριμένο, κοιτάξαμε το γράμμα του άρθρου 16 και συγκαλέσαμε μια επιτροπή που λέγεται Μικτή Επιτροπή Joint Committee. Συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα και την αρχή της επόμενης εβδομάδας και στις 16 και 17 Μαρτίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και θα συζητηθεί το θέμα εκεί και ενδεχομένως, ενδεχομένως δεν θέλω να προεξοφλήσω τίποτα, τότε να ληφθεί κάποιο μέτρο από πλευράς του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν θέλω να το προεξοφλήσω, ας περιμένουμε τη διαδικασία. Ένα τελευταίο, <laughs> λέει για τρίτη φορά ο μιλητής και διακόπτει ο πρόεδρος. Ε, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία ζημία ούτε ηλική ούτε οικονομική και το ελεγκτικό συνέδριο έχει επιβεβαιώσει στον οργανισμό μας ότι είναι εντάξει τα οικονομικά και οι λογαριασμοί και αυτό θα παρακαλούσαμε να χορηγήσετε την απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Um, Για να κλείσουμε θα ξαναδώσω το λόγο στον Σενάφο Σταυρακάκη. Συμφωνώ και εγώ με αυτό που πριν ο Σενάφο Στάς. Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε σήμερα απαιτεί περαιτέρω εμβάθυνση. Θα το βάλουμε στην ημέρηση διάταξη με επόμενη συνεδρίαση. Όλα τα θέματα αυτά που σήμερα το πρωί εθίχθησαν και άλλα επειδή δεν είχαμε χρόνο για σήμερα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις πολύ επικοδοποιητικές παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ επίσης θερμά τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Σουσέα ότι θα συνταχθεί μελέτη δικτών έτσι ώστε να βοηθήσει την Επιτροπή μας ε, στην περαιτέρω αξιολόγηση ε, των οργανισμών. Ε, αυτό που μόλις τώρα ανακοινώσετε ότι σε επόμενη ημερήσια διάταξη θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα με καλύπτει απολύτως και επομένως δεν έχω να αναφέρω τίποτα παραπάνω εφόσον θα συζητηθούν στην Επιτροπή μας. Σε κάθε συζήτηση που γίνεται όσον αφορά την απαλλαγή ε, νομίζω ότι δίνεται η ευκαιρία να τονιστούν ορισμένα πράγματα αλλά όπως υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους ε, ο ακριβής ρόλος αυτής της συζήτησης είναι η δημοσιονομική διαφάνεια και η απαλλαγή ή όχι των οργανισμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σα θυμίζω ότι προθεσμοί για τι τροπολογίε 8 Μαρτίου, 12 η ώρα. Τώρα αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Αρχίζει η συνεδρίαση των συντονιστών. Καλώ του άλλου ε, συναδέλφου, τους, τους αποχαιρετάω ε, ήδη από τώρα, μπορείτε να φύγετε.